Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ακούσουμε τις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κατάσταση στη Βουλγαρία. Δείχνω, δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Λεσκεβίτσους. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, αντιπρόεδρε τη Επιτροπής. Είμαι ενθουσιασμένος που στέκομαι ενώπιόν σα. και θα είμαι συχνός προσκεκλημένος σας 179 μέρες. Προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Αξιότιμοι βουλευτές, ζητήσατε να κάνω μία δήλωση για την τωρινή κατάσταση στη Βουλγαρία. Αυτή η κατάσταση ε, οδήγησε σε ε, σοβαρές ανησυχίες σε όλο το πολιτικό φάσμα του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω ότι πολιτικός πώς είναι αρκετά σοβαρό το θέμα ώστε να γίνει μια σχετική συζήτηση και σας ευχαριστώ που την οργανώσατε σήμερα. Θα ε, θέλαμε λοιπόν ε, να διαβιβάσουμε τις απόψεις του Συμβουλίου αλλά δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να το κάνω γιατί το Συμβουλίο δεν έχει συζητήσει την ε, χώρια κατάσταση στη Βουλγαρία και δεν έχει τίποτα να πει για αυτό το θέμα. Είναι σπάνιο εξάλλου να διεξαγόνται τέτοιε συζητήσει για την χώρια κατάσταση κρατών μελών στο Συμβούλιο. Όμως η κατάσταση διαφέρει για το Κοινοβούλιο όπως και για, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό αλλά και για όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Συζητούν ζητήματα δημοσίου κοινού ενδιαφέροντος. Ο δικός μου ρόλος είναι να εκπροσωπώ το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο δικός σας. Εκπροσωπούμε 28 κράτη-μέλη, εκ των οποίων η Βουλγαρία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις για το ζήτημα. Δεν είναι απλό να εκπροσωπεί κανείς το Συμβούλιο. Όταν μπορεί, ε, κοινοποιεί τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, αλλά λειτουργεί και ως διάβλος ε, αντίστροφης ροής πληροφοριών. Με ιδιαίτερη προσοχή θα διαβοβάσω το περιεχόμενο των σημερινών μας συζήτησεων και ε, σίγουρα θα εκφραστούν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα σήμερα, τις οποίες και θα διαβιβάσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Παρόλα, Η Επίτροπος, κυρία Ρέντινγκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή εξέτασε τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βουλγαρία και βεβαίως ε, σεβόμαστε τις εθνικές αρμοδιότητες. Ορισμένες όμως καταστάσεις μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αναφέρομαι ε, στο θέμα της, ε, του φορέα των μυστικών υπηρεσιών και του επικεφαλής αυτού που θα πρέπει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Η Επιτροπή καλωσορίζει και δέχεται το γεγονός ότι το, Ευρωπαϊκό, το ε, Βουλγαρικό Κοινοβούλιο ήρε αυτό το διφορούμενο. Όταν ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ε, διασαφήνισε αυτό το ζήτημα. Μιλήσαμε για τις ανησυχίες όχι μόνο της Επιτροπής, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών της Βουλγαρίας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τους μελλοντικούς διορισμούς σε στρατηγικές θέσεις με βάση την αξιοκρατία των υποψηφίων. Τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα και οι διαδηλώσεις στη Βουλγαρία καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία από την βουλγαρική κοινωνία για την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Η Βουλγαρία θα πρέπει να συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις και να ε, αναμορφώσει το, τον δικαστικό τομέα και να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς επαλήθευσης και ελέγχου για την περίπτωση και της Βουλγαρίας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη πληρούν τις υποχρεώσεις τους και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ε, βοηθά την Βουλγαρία για να αποδώσει στις μεταρρυθμίσεις της μέσω του μηχανισμού ε, επαληθεύσεων και ελέγχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ο κύριος Βέμπερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κυρία Τη Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει σε πώς να δούμε εδώ ποιος από τους σοσιαλιστές είναι παρόν για να μιλήσει για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν φύγει όλοι. Αλλά όταν μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό θα πρέπει να μας αφορά σε όλες τις χώρες και στη Βουλγαρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ε, πήρα καμία απάντηση. Λίγοι σοσιαλιστές έχουν παραμείνει στην αίθουσα, ίσως κάποιος να μου δώσει κάποια απάντηση. Ο Χανές Φόμποντα θα μας πει εδώ βεβαίως ότι θα αναγκαστούμε να καταπιούμε κάποιες από αυτές τις παραβιάσεις. Αυτό είναι κάτι που το είπε λίγο πολύ ο Χάνες Φόμποτα. Με ποιο τρόπο, αν θέλετε, οι ψηφοφόροι δεν υποστήριξαν σε πλειοψηφία τους σοσιαλιστές και παρόλο που υπήρξε υπόσχεση για υποστήριξη από μέρους των Ρώσων, αναρωτιόμαστε τι συνέβη στη Βουλγαρία. Έχει δίκιο η Επίτροπος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ότι είναι δραματική η κατάσταση, ότι υπάρχει διαφορά, οργανωμένο έγκλημα και κανένας, απολύτως κανένας κοινοβουλευτικός έλεγχος. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Οι εκπρόσωποι των ε, μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης παίζουν ένα ρόλο που δεν είναι ρόλος καθόλου αρμόζουν σε επικεφαλής ομάδων επιρροής και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι αυτό καμία σωστή αντίληψη της δημοκρατίας και ελπίζω να το καταλάβουν αυτό οι σοσιαλιστές και να λογικευτούν σε αυτά που λένε. Πραγματικά θα πρέπει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση έτσι ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα του ανθρώπου να μην παραβιάζονται στη Βουλγαρία. Θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω από όλους εδώ τους πολιτικούς φίλους των σοσιαλιστών στην Βουλγαρία να πούν την αλήθεια, να δεχτούν την αλήθεια, γιατί αυτό που μας αφορά και μας ενδιαφέρει εδώ είναι να υπάρξει μια πραγματική δημοκρατία και σταθερότητα στην Βουλγαρία. Κύριε Βεν, δέχεστε μια ερώτηση, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κύριλοφ. Κύριε Βέμπερ, Εσείς ήσασταν ο εκπρόσωπο του κόμματος Γκέρμπεδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρουσία του κόμματο σας ε, στο Κοινοβούλιο ε, είναι η ακόμη και από αυτή των σοσιαλιστών. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους συναδέλφους σας. Κάνετε μάλλον γενικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Το αν κάποιος εδρεύει όχι στο κοινοβούλιο, τι σχέση έχει με την πολιτική υποστήριξη. Μέλη του ΑΤΑΚΑ ποτέ δεν μας ε, ψήφισαν ε, διαφοροποιείται την εγγραφή σε κάποιο κόμμα με την ε, ε, πολιτική υποστήριξη εδώ στο Κοινοβούλιο. Εμείς προσπαθήσαμε ε, να επανέλθουν οι σοσιαλιστές στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ από τις τρεις. Συζήτησα όλο το θέμα της Ουγγαρίας και αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι οι σημαντικοί ομιλητές από μέρους των σοσιαλιστών φύγαν. Όλοι, όλοι. Δεν υπάρχει κανείς. Έφυγε και ο Φερχόστατ, έφυγε και ο Κονβεντίτ. Αυτό που επικρίνουμε είναι ακριβώς αυτό, την μονομέρεια. Οι σοσιαλιστές δεν έχουν την δύναμη και το θάρρος να πούν την αλήθεια στους φίλους τους στη Βουλγαρία και να δεχτούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Ξέρουμε σήμερα ποιο είναι ο ρόλος των σοσιαλιστών στη Βουλγαρία. Έχουν συνάψει συμφωνία με τον διάβολο. Κύριε Βέμπερ και άλλη μπλε κάρτα. Η κυρία Γιώτοβα. Παρακαλώ. Βέμπερ, колкото повече ви слушам, άκουσα με προσοχή. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν είστε σίγουρος σε σχέση με τις αρχές σας. Γιατί άλλαξε ο λόγος σας τώρα που μιλάμε για τη Βουλγαρία σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση για την Ουγγαρία. Μήπως ακολουθείτε οδηγίες, εντολές, ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, ερώτηση. Ήταν δίκαιες οι εκλογές που ανέδειξαν την τωρινή κυβέρνηση στη Βουλγαρία. Για ποιο λόγο ζητάτε εσείς προώρες εκλογές. Δηλαδή αν έρθω εγώ στην πατρίδα σας και ζητήσω προώρες εκλογές το βρίσκεται θεμητό. Κοιτάξτε, αν θέλετε εδώ να συγκρίνουμε με την κατάσταση στην Ουγγαρία, μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει μία συμμαχία, όπως έκανε ο Βίκτορ Όρμπαν, με τους ακροδεξιούς. Αυτό θα ήταν το αντίστοιχο. Και το κόμμα Ατάκα. Είστε πραγματικά στο όριο και τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να λογικευτείτε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Ο κ. Μωράης, για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Βέμπερ, επειδή ο κύριος Ντόλ δεν είναι παρόν και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους παίχτες, ε, όπως τον κύριο Κονβεντίτ, ο οποίος δεν, ήταν, ε, δεν είναι σοσιαλιστής από όσο γνωρίζω, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Είχαμε τη συζήτηση αυτή για την Ουγγαρία και μιλήσαμε για συστηματικές αλλαγές του συντάγματος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως το θέμα που μας απασχολεί στη Βουλγαρία είναι πολύ διαφορετικό, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ανησυχίες για τη χρήση των μεταρρυθμίσεων και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Στη Βουλγαρία έχουμε ε, τον λάθος άνθρωπο σε μία στρατηγική θέση και μία αναδιοργάνωση ε, του φορέα αυτού, του οργανισμού αυτού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, δυστυχώς δυσλειτουργεί και δεν συνεργάζεται και με τις ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές όπως θα έπρεπε. Ε, θα μπορούσε να αναχαιτήσει την ε, καλή συνεργασία με τη Βουλγαρία ως προς τον ε, μηχανισμό ελέγχων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τις ε, θεσμικές εξελίξεις και να διευρύνουμε το πλαίσιο διερεύνησης και του σκανδάλου υποκλοπών. Θα ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό προτείναμε, όπως και στην Ουγγαρία, να υπάρχει ένας μηχανισμός εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να ε, καταπραίνουμε και τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο κύριος Βέμπερ. Και αυτή είναι απάντηση από την ομάδα μας. Κύριε Μωράης, δεχόσαστε μία μπλε κάρτα. Έχω και την επιλογή. Ο κύριος Στογιάννοφ. Σε σχέση με κάτι που προείπατε κύριε Μωράης και που σχετίζεται με την ε, ανάμιξη ε, συμμετοχών και την ε, τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού. Εσείς πιστεύετε ότι ο οργανισμός είναι μια νέα στάση? Δεν ξέρω ποιον ακούγατε, πάντως όχι εμένα. Είπα ότι ο, το, ο λάθος άνθρωπος βρίσκεται σε λάθος θέση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζεται μία επαναδιοργάνωση αυτού του οργανισμού για να μπορέσει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είπα. Και αυτό ξαναλέω. Από τους φιλελεύθερους, η Σμενόβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η, πιστο... η χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει αναστάτωση στη μισή Ευρώπη τουλάχιστον και η περίπτωση της Βουλγαρίας δεν διαφέρει, αλλά σε αντίθεση με την συζήτηση που είχαμε πριν, στη Βουλγαρία λειτουργεί ο νόμος θεσμικά η Βουλγαρία επέλεξε τη δημοκρατία, έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, υπάρχει το κοινοβούλιο που είναι δραστήριο. Αν και ε, πολλοί δεν το αποδέχονται αυτό και υπάρχουν και οι δημόσιες ε, διαδηλώσεις που είναι δημοκρατικές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ανταποκριθεί. Το κόμμα αυτό στο οποίο προναφέρθηκε ο κύριος Βέμπερ ε, δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση, δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση και για αυτό ε, στην περίπτωση της ΑΤΑΚΑ δεν υπάρχει συμμετοχή και το ΕΛΚ όταν ανέκεψε το ζήτημα αρχικά δεν είπε τίποτα. Η κυβέρνηση σήμερα αποτελεί μια ε, επικοδομητική εναλλακτική λύση και θα πρέπει να της δοθεί μια ευκαιρία να σταθεροποιήσει τη χώρα μέσα στα πλαίσια ενός νέου προγραμματισμού για την προετοιμασία των εκλογών. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι πρωταρχικό ε, το κράτος δικαίου. Κύριε Γουσμάνα, δέχεστε μπλε κάρτα. Ο κύριος Κόβατσεφ. Κυρία Ισμάνοβα, δύο ερωτήσεις ε, θα ήθελα να σας κάνω. Με ναι ή όχι μπορείτε να απαντήσετε. Η τωρινή κυβέρνηση του κυρίου Ρισάσκη παραβιάζει τα δικαιώματα ναι ή όχι και η εκστρατεία για την οποία μιλήσατε όντως είναι δημοκρατική ναι ή όχι. Δεν θέλω να μου δώσετε μακρόσκελη απάντηση. Ένα ναι ή όχι. Κύριε Κοβάτσεφ, ε, ξέρετε, η Η τωρινή κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη αν δεν είχαν γίνει αυτές οι εκλογές. Και εξάλλου αυτά που έκανε το κόμμα σας σε εκλογές θα θυμούνται όλοι. Ευχαριστώ κύριο Σταβάρης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή μετά την Ουγγαρία περνάμε στη Βουλγαρία και βλέπουμε τη νέα κρίση με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προσεχή χρόνια. Την κρίση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολύ βαθύτατη μάλιστα σε σχέση με την οικονομική κρίση, το ξέρουμε από την παρελθούσα εμπειρία μας. Ε, είδαμε εκλογές που μπορεί κανείς να αμφισβητήσει σε μεγάλο βαθμό ως προς τη δικαιοσύνη τους ε, στη Βουλγαρία όπως και στην Ουγγαρία. Ε, έχουμε λοιπόν έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία που επέστρεψε στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα έχουμε τους νέους Βούλγαρους που όπως οι νέοι σε όλη την Ευρώπη θέλουν μία χώρα που δεν επικρατεί η διαφθόρα και όπου γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Δεν μπορούμε να περιέλθουμε σε μία κατάσταση όπου είναι ανίσχυρες οι δημόσιες αρχές λόγω αυτής της κατάστασης ε, και γι' αυτό προτείνεται να συστηθεί η Επιτροπή της Κοπενχάγης ούτως ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα των εθνικών νομοθεσιών με το άρθρο 2 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι κρούεται και ο κόδωνας κινδύνου μέσα στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής, ε, δηλαδή μεταβαίνουν ε, κλιμάκια στην ελόγω χώρο για να ελέγξουν την κατάσταση σε κάθε χώρα. Στην Βουλγαρία, στην Ουγγαρία και σε οποιοδήποτε χώρο ο στόχος είναι να υπερασπιστούμε τα ε, οικομενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Καλά, ευχαριστούμε κύριε Ταβάρης. Ο κύριος Μέρφη τώρα ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Βουλγαρία είναι άλλη μια χώρα που μπαίνει στον παγκόσμιο αγώνα κατά της ευτόχειας της ε, και της διαφθοράς. Ε, βλέπουμε ότι όλοι είμαστε ενωμένοι, η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Βραζιλία με τα λαϊκά συλλαλητήρια κατά ε, των κυβερνήσεων, διότι τους ζητούμε να εργάζονται για εμάς. Ε, και αυτό εκφράζει το, η λαϊκή οργή κατά της ε, τάξη. τάξης. είναι υποκριτικό από πλευρά των κομμάτων να κατηγορούν οι μεν τους δε για την μιζέρια και την φτώχεια των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι για τη δημιουργία της. Είναι η φτωχότερη ε, χώρα η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κάτω από 100 ευρώ οι συντάξεις, ε, κάτω από 400 ευρώ η βασική μισθή και μέσα σε αυτή τη φτώχεια γίνονται οι αποκρατικοποιήσεις. Είναι δεινή η κοινωνική κατάσταση και ταυτόχρονα η εργατική τάξη είναι αυτή που πρέπει μέσα από τα συνδικάτα να αγωνιστεί, να οργανωθεί, ούτως ώστε μέσα από τον αγώνα να γίνουν ζωσπαστικέ αλλαγέ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μέρφυ, ο κύριο Μπίνεφ. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε σήμερα Βούλγαρου στο δρόμο. Διαμαρτύρονται, διαδηλώνουν γιατί έχουν την ελευθερία να το κάνουν. Στο παρελθόν η κυβέρνηση, εάν ε, τολμούσαν να εκφραστούν κατά της ε, κυβερνητικής πολιτικής, τους περιόριζε και τους συνελάμβανε. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αντιπολίτευση και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καλούμε δημοκρατικό κόμμα αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά επιθυμούν να οδηγήσουν την Βουλγαρία στην απόγνωση και στη φτώχεια. Γιατί τους ε, υποστηρίζετε, γιατί στηρίζετε τον Σρετάνοφ, τον Βούλγαρο Καντάφη και τις ε, δυνάμεις αυτές οι οποίες υποστηρίζουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι Είμαι πολύ περήφανος γιατί πρώτη φορά εκατοντάδες χιλιάδες νέοι στην χώρα μου βρίσκονται στους δρόμους και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των πολιτών. Τι είναι αυτό που τους έφερε στο δρόμο και τους οδήγησε στο να διαδηλώσουν. Είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις κατηγορίες που ακούμε εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Το βασικό πρόβλημα κυρίες και κύριοι στην Βουλγαρία είναι ότι πριν από τέσσερα χρόνια αυτά τα κόμματα τα οποία σήμερα είναι στην κυβέρνηση ήταν άσπονδοι εχθροί. Σήμερα σε μια πολύ αφύσικη και τελείως παράλογη συμμαχία δημιούργησαν κυβέρνηση. Ο μόνος δημοκρατικός τρόπος να βγούμε από αυτό το διέξοδο είναι να γίνουν νέες εκλογές. Δίας μέρα. Ο κύριος ε, Μπορισόφ έκαναν, ε, έκανε μια πολύ σοβαρή εργασία για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς. Η νυν κυβέρνηση θέτει επικεφαλής της ΣΑΝΣ που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ε, βάζει η πάγη της ΣΑΝΣ στην αστυνομία. Με ποιο στόχο για να ε, υπάρξει σκοταδισμός και απόκρυψη. Και συμμερίζομαι αυτά που είπε ο κύριος Μωράης, ο οποίος πολύ ισορροπημένα εξέφρασε τις ανησυχίες του για αυτό τον διορισμό του Ελέιαν Πένσκι και δέχομαι αυτές τις ανησυχίες που εξέφρασε και η Επίτροπος η κυρία Ρέντινγκ. Τα στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά στα πλαίσια της ασφάλειας στη Βουλγαρία. Μιλάμε για μία υπηρεσία που είναι πολύ ευάλωτη και αυτό θα μπορούσε να σταθεί ολέθριο για την ασφάλεια της χώρας. Άρα η Συμμαχία για τη Σοσιαλιστική Βουλγαρία, δηλαδή το 26,5% συν την ΑΤΑΚΑ 7,35% μας δίνουν αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Δηλαδή το 7,35% είναι αυτό το οποίο αποφασίζει στη Βουλγαρία. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Διαστεμέρα. Ο κύριος Λόπες Αγγιγιάρ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ορισμένα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια των ε, πολιτικών ελευθεριών συμμετείχαμε στην προγενέστερη κατάσταση, ε, συζήτηση με συγχωρείτε, ως προς την κατάσταση ε, στην Ουγγαρία και μιλήσαμε, μιλάμε τώρα και για την κατάσταση τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν ε, κοινά σημεία και δεν υπάρχουν δύο μέτρα και στάθμα λυπούμεθα, διότι αυτή η συζήτηση αντί να προβάλλει το, την ευρωπαϊκή θεώρηση, οδηγεί σε μία σειρά εθνικών αντιφάσεων θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανησυχούμε πράγματι για αυτή την υπηρεσία εθνικής ασφάλειας όπου έγινε ένας διορισμός απαράδεκτος. Έχουμε λόγους ανησυχίας για αυτές τις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στη Βουλγαρία που δείχνουν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θεμελιώδη δικαιώματα εκεί όπου υπάρχουν παραβιάσεις έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και την τήρηση του κράτους δικαίου όπως μιλήσαμε και το 2012 για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο κύριος Πίρκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Η σημερινή κυβέρνηση σοσιαλιστική στη Βουλγαρία μετά τις εκλογές και την επιλογή προσώπων για πολύ σημαντικές θέσεις βρίσκεται σε μια πάρα πολύ απογοητευτική κατάσταση. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πρώτον, το θέμα των αρμοδιοτήτων, των ε, υπηρεσιών αυτών, που έχουν αρμοδιότητες για θέματα ασφάλειας. Πρόκειται για ανεξέλεγκτες υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά δεν ελέγχονται και δεν υπόκεινται σε κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη λοιπόν δραστηριότητα για τους επικεφαλείς αυτών των υπηρεσιών, κύριε Μπέσκι Υπάρχουν εντολές χωρίς περιορισμούς και αυτά πραγματικά είναι πρωτοφανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άνθρωποι με τέτοιες αρμοδιότητες, με τέτοιες δεξιότητες και προσόντα να αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις. Και θα πρέπει η Επιτροπή πολύ προσεκτικά να εξετάσει αυτή την περίπτωση στη Βουλγαρία. Ευχαριστώ κύριος Κάλφιν, λέει η Πρόεδρος, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να μην υπάρξει καμία παρανόηση θα σας έλεγα ότι είναι ξένοφοβικό, εθνικιστικό, ακροδεξιό κόμμα το ΑΤΑΚΑ που πόρο απέχει από τις ευρωπαϊκές αξίες. Η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Μπορίσοφ ε, υπολόγιζε στις ψήφους του ΑΤΑΚΑ. Το ίδιο ισχύει και στη σημερινή κυβέρνηση. Αλλά τώρα ε, το να αφαιρέσουμε από τον ΑΤΑΚΑ το καταλητικό του ρόλο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε και τον ΚΕΡΠ. Γιατί άμα τον ΚΕΡΠ πάει στο κοινοβούλιο θα αποκλειστεί το ΑΤΑΚΑ. Ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών μίλησε προσωπικά με τον κύριο Μπόρισοφ, του ζήτησαν να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο. Αυτός και τον Γκέρμπε, εσείς τι θα λέγατε. Ευχαριστούμε, θα ακούσουμε τον κύριο Γκάλερ για την απάντηση. Θα μιλήσω ε, αγγλικά. Ε, κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα στη Βουλγαρία είναι ότι γίνεται από την παλιά νομενκλατούρα μία τελευταία απόπειρα και μιλώ εδώ και για την ολιγαρχία και για τα ρωσικά συμφέροντα και για τους σοσιαλδημοκράτες να αναστρέψουν την τάση προτού μπορέσουν να παγιωθούν δημοκρατικά θεσμικά όργανα βάσει του συντάγματος. Ο, ο, ο πρώην Πρωθυπουργός Βιγγέννη θέλει να επαναφέρει τον κύριο Δημήτρη και να γίνει γενικό γραμματέα ε, του Υπουργείου Εξωτερικών. Γνωρίζετε το ρόλο του στο πρώην κομμουνιστικό ε, Καθεστώ. και παρότι είναι εξαιρετική συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη και συνεργάστηκαν για την καταπολέμηση τη οργανωμένη εγκληματικότητα. Αυτό έθεσε εν κινδύνο την ολιγαρχική τάξη και γι' αυτό ε, με αυτό το το κανάλι 7 είχε τόσο κέριο ρόλο για την καταγγελία της νοθείας στις εκλογές ο κύριος Κυριλόφ. Έπρεπε να ανταμυφθεί και ο κύριος Στάνης, εφόσον σοσιαλιστής ε, ηγέτης, ε, είναι αυτός που συντονίζει αυτή τη δράση. Καλό θα, καλά θα κάνατε να έχετε μια ομή και ειλικρινή συζήτηση μαζί του. Ο κύριος Τσβέρ για όλα αυτά τα πάρα πολύ ευαίσθητα και λεπτά θέματα που αφορούν τη μεταβατική περίοδο σε αυτές τις χώρες. Ο εκδημοκρατισμός δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και τα δημοκρατικά κόμματα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι σοσιαλιστές. Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε την ε, κυβέρνηση και παρόμοιες καταστάσεις ζήσαμε και στη Σλοβενία. Είχαμε δύο επιτυχημένες ε, και νόμιμες κυβερνήσεις και το παράδοξο είναι ότι το Σλοβενικό κόμμα SDS και το GERP είναι αυτοί που έχουν αναλάβει την προσπάθεια και τη μάχη κατά της διαφθοράς. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενδυναμωθεί το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε κάθε συζήτηση που έχουμε ε, εισάγονται πολλά και σημαντικά ζητήματα και χαίρομαι διότι ε, προτάθηκε αυτό το θέμα και εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη. Αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη τα πραγματικά γεγονότα, διότι έχουν ακουστεί πολλά και αντιφατικά. Στη Βουλγαρία το ε, βασικό πολιτικό κόμμα ε, δεν ε, έλαβε πλειοψηφία και γι' αυτό έπρεπε να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού και πολλοί για να εκφράσουν την ε, δυσαρέσκειά τους δεν προσέρχονται στην εργασία, ούτε στο κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση στη Βουλγαρία ε, θα πρέπει να έχει μια, τη δυνατότητα να μπορέσει να δράσει. Μάλινοφ, αγαπητοί συνάδελφοι, τα πολιτικά γεγονότα στη χώρα μου συζητήθηκαν ε, στο σώμα αυτό και αυτό τον καιρό είχαμε πολλές διαδηλώσεις στη Βουλγαρία, πρόορες εκλογές, μια νέα κυβέρνηση, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και πάλι πρόορες εκλογές. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τους πολιτικούς. Και τώρα λοιπόν στρέφονται στην Ευρώπη γιατί θέλουν ε, να μάθουν τι γνώμη έχουν οι ομότιμοι πολιτικοί. Από ό,τι διαπιστώνω εδώ φαίνεται ότι έχουν πολύ καλούς λόγους να μην εμπιστεύονται ε, ούτε, ούτε τους Ευρωπαίους πολιτικούς και με κάθε ειλικρίνεια θα υπάρξει περισσότερος ε, ευρωσκεπτικισμός και ε, θα αναζωπυρώνεται οι εθνικισμοί. Γιατί ε, θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα όταν ε, κρίνουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλουμε το καλό τη πλειοψηφία και το σεβόμαστε γιατί εκείνοι αποφάσισαν να οργανώσουν τη σημερινή συζήτηση και γίνονται σεβαστές οι αρχέ της δημοκρατίας. Όμως υπάρχει σοβαρό έλλειμμα αλήθειας σε αυτή τη συζήτηση. Εξαιτία του Γκέρμπ και των οπαδών του. Ήταν καταστροφικά τα αποτελέσματα της κυβέρνησης ε, Γκέρμπ και τότε δεν συζητήθηκε το ζήτημα καθόλου εδώ στο Κοινοβούλιο. Τώρα που αποχώρησε το Γκέρμπ το συζητάμε. Και ακούμε εδώ ότι έπρεπε να επιστρέψουν στην κυβέρνηση κύριοι όπως ο κύριος Μπόικο Μπόρισοφ. Μα καταψήφισε ο λαός ε, το Γκέρμπ μετά από 3,5 χρόνια, μετά από μια ανεπιτυχή κυβέρνηση που δεν κατάφερε να εξασφαλίσετε καν δίκαιες εκλογές. Με τόσα σκάνδαλα Πώς μπορείτε αγαπητοί συνάδελφοι να υποστηρίζετε ακόμη το Γκέρμπε και τους οπαδούς του. Ευχαριστούμε. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς η κυρία Λούπτσεβα δεν ήταν νωρίτερα εδώ για να ακούσει την συζήτηση πριν από μερικά χρόνια που ξεκίνησε εδώ κατά της κυβέρνησης Γκέρμπ. Ευτυχώς, ευτυχώς, οι πολίτες στη Βουλγαρία δεν ψήφισαν όμως το κόμμα αυτό που σήμερα βρίσκεται στην κυβέρνηση μαζί με το κόμμα Ατάκα. Γιατί λοιπόν δεν κάνετε τίποτα κατά του Ατάκα, απάντηση. Για τους Βούλγαρους νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Εκτός του Γκέρμπ που μποϊκοτάρει τη συμμετοχή στο Κοινοβούλιο. Βλέπετε ότι οι υπόλοιποι στηρίζουν την κυβέρνηση. Η Ατάκα δεν υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση και όλοι το ξέρουν γιατί δεν είναι υπέρ της ε, καταπολέμησης της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Μιλούμε για διπλά standards εδώ, για διπλά πρότυπα. Και πραγματικά πρόκειται για κάτι που όπως και η κυβέρνηση Μπόρισοφ σε τακτική βάση έκανε προσπάθειες. Σήμερα βλέπουμε ότι η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να ενδυναμώσει την ασφάλεια, κάτι που δημιουργεί ανησυχίες. Αυτό που συνέβη στο παρελθόν με την προηγούμενη κυβέρνηση είναι να υπάρχει εκβιασμός κατά των επιχειρήσεων, εκβιασμός τους επιχειρηματίες. Και το ΕΛΚ βεβαίως είναι κατά αυτών των προτάσεων. Πώς είναι δυνατόν. Σήμερα μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει αναλάβει πριν από ένα μήνα και προσπαθεί να επαναφέρει τη Βουλγαρία πίσω στην δημοκρατία. Η κυρία Ρέντινγκ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί σε σχέση με τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία και το ίδιο και για τα κράτη-μέλη. Δεν θα ε, διστάσουμε αν διαπιστωθεί παραβίαση των βασικών νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σοβαρή παραβίαση των ε, ευρωπαϊκών αξιών, να δράσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ακούσει τα ίδια πράγματα πολλές φορές. Και σας το ξαναείπα όταν μιλούσαμε για την Ουγγαρία φέτος, πέρσι, θα είμαστε σε εγρήγορση. Όπως έχουμε ήδη πράξει στο παρελθόν, αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι ε, είναι πολλωμένο το πολιτικό κλίμα στην ε, Βουλγαρία και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Βουλγαρίας ε, για να καταλήξουν σε μια συνενετική λύση ώστε να επικρατήσει και ευημερία και σταθερότητα στη χώρα. Πρόεδρε, οι δύο συζητήσεις ε, που έκανε σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο δείχνουν πόσο σημαντικό είναι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να προαγάγουν το κράτος ε, δικαίου. Κάποια όργανα τα έχουμε στη διάθεσή μας, συνεργασία και ο μηχανισμός επαλήθευσης, Φερρυπίν, και μπορούμε να αντλήσουμε τα διδάγματα μας από τη χρήση αυτών των μηχανισμών. Όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα που έχουμε για να απαντούμε ε, σε ε, καταγγελίες ως προς ε, το κράτος δικαίου και το αν γίνεται σεβαστό. Αυτά σας είπα και στη συζήτηση που κάναμε για την Ουγγαρία. Όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν τον πολιτικό διάλογο για αυτά τα ζητήματα. Επίσης συνεχίζει το διάλογο με τις δικαστικές αρχές διότι είναι προς συμφέρον όλων και κυρίως των πολιτών της Ένωσης που αναμένουν σημαίνουν ε, προστασία των ε, θεμελιωδών αξιών και των δικαιωμάτων τους. Ε, σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, και εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος Λέσκεβίτσους. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. and good note Άκουσα με προσοχή την ε, συζήτηση και είδαμε ολόκληρο το φάσμα των ε, παραβιάζων ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ εκπροσωπώ το Συμβουλίο και δεν αρμόζει ως εκ τούτου να δώσω συγκεκριμένε απαντήσει ε, για τη σειρά αυτών των ανησυχιών που εκφράστηκαν για την ε, τωρινή πολιτική κατάσταση στη Βουλγαρία. Πολλοί από εσά όμως ε, ξεκαθάρισαν ότι έχουν τι ανησυχίε για τι πρόσφατες πολιτικέ εξελίξει και θα σα κάνω μία αναφορά και θα διαβιβάσω τα σχόλιά σας στους συναδέλφους του Συμβουλίου ε, για όλη τη σημερινή συζήτηση και θα επανέλθω με τα σχόλιά τους. Βάσει του άρθρου 216 παράγραφο 4 σα ενημερώνω ότι δεν έχουν ζητηθεί να ψηφιστεί το διορθωτικό το οποίο αναγγέλθηκε σε 17 και 30. Το διορθωτικό λοιπόν θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Προχωρούμε τώρα στην ε, δήλωση της Επιτροπής